Εν τω μεταξύ να σα πω ότι έχουμε κοινή συνεδρίαση τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για να ψηφίσουμε για την ε, προσωρινή συμφωνία που προέκυψε τον τρομερή διάλογο για την νομοθεσία για τον έλεγχο ροών που εισέρχονται ή εξέρχονται τη Ένωση, Ρεντελβό και Λόπες Αγγιλάρ. Οι επιτυχής ε, ο τριμερής διάλογος. Δεν ξέρω αν θέλουν κάτι να πούν οι εισηγητές. Έχουν το δικαίωμα. Ο Χουάν Φερνάντο βλέπω. Τουλάχιστον να ευχαριστήσω την κυρία Ντελβό, ε, το επιτελείο μας και τους συναδέλφους που είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης μετά τις ε, μακροσκελείς διαπραγματεύσεις θέλαμε να δείξουμε ότι κατανοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο ε, σημαντικό είναι ο έλεγχο ε, του ρευστού στα σύνορα με αναλογικό τρόπο και με σεβασμό προ τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάνω απ' όλα στην κυρία Ντελβό για την ε, συνεργασία που καταφέραμε να πετύχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ωραία. Καλά κάνετε και μεταφέρετε αυτές τις ευχαριστίες γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ε, διοργανικής συνεργασίας αλλά και μεταξύ των επιτροπών. Η ισχύ εν λοιπόν πετύχαμε πολλά θετικά αποτελέσματα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Ωραία, ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφορία, για τη δοκιμαστική ψηφορία πάντα. Πέρας. Ωραία, για το συμπεφωνημένο κείμενο στο πλαίσιο της διοργανικής διαπραγματεύσης με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. 68 υπέρ, Μηδέν. κατά, τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια. To the two co-rapporteurs and to uh, all the shadows and the staff secretariat and negotiating team. Thank you. Liebe colleagues, now we move back. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Επιστρέφουμε στις ψηφοφορίες εικόνων. They have to make some new re... re... Η δερμηνία θα σταματήσει τώρα. Καλό σας βράδυ.